Φεβρουαρίου 2014. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί τη 6η Φεβρουαρίου πάντα διατίθενται. Έχετε αντιρρήσει, ενστάσει ω προ τα αυτά. Όχι, τότε θεωρείται εγκεκριμένο το συνοπτικό πρακτικό.